θα ήθελα να κάνω μια επίσημη ανακοίνωση. Πιο συγκεκριμένα, η σύσταση για απόφαση που ε, υπέβαλε η Επιτροπή Οικονομικών ε, και Νομισματικών Υποθέσεων να μην υπάρξει αντίρρηση σε πράξη κατεξουσιοδότηση που ανακοινώθηκε χθε. Δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις ε, μέχρι τώρα και βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 6 του κανονισμού η σύσταση λοιπόν εγκρίνεται. Θα δημοσιευθεί με την έγκριση των πρακτικών αύριο 5η 9 2016.